Άρχεται τη συνεδρία, κυρίε και κύριοι. Καλημέρα σα. Πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Συμβουλίου για την νομική βάση του μηχανισμού αξιολόγηση τη Συμφωνία του Σέγγεν. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία οφθαλμοσύλληψης catch the eye κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Äh, Κύριε Φερχόφστατ, μπορείτε να ηρεμήσετε. Ε, μπορείτε να κάνετε μετά τις ε, έντονες ε, δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Μπότσκοφ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζω την κυρία Μάλμστρομ επίσης. Έχουμε συμφωνήσει ότι η κυρία Μάλμστρομ θα λάβει το λόγο μετά από τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων για τη δική της δήλωση. Οπότε το λόγο έχει η Προεδρία του Συμβουλίου με τον κύριο Μπότσκοφ. Σας δίνω το λόγο κύριε Μπότσκοφ. formand for Europaparlamentet, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να πάρουμε το λόγο με αφορμή τη συζήτηση αυτού του ιδιαίτερου σημαντικού θέματος.